θα επιτρέψει την... Ε, θα επιτρέψει επίσης την προώθηση του ευρωπαϊκού δικαίου και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Έκλεισε η συζήτηση. Αύριο στις 12.30 θα υπάρξει ψηφοφορία και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για την έκθεση του Λουίτζι Μπερλιγκουέρ, διαδικασία της Μπολόνια για τέσσερα λεπτά λεπτά έχει το λόγο Πρόεδρε, ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι η πρωτοβουλία για τη διαδικασία της Μπολόνια. Έχοντας κατά νου ένα σημαντικό στόχο. Ότι δηλαδή τα πτυχία που αποκτώνται σε ευρωπαϊκό έδαφος θα πρέπει να έχουν γενικότερη αξία. Εάν κανείς λάβει ένα τίτλο, ένα πτυχίο σε ένα κράτος μέλος, θα πρέπει όλα τα άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης να τον αναγνωρίζουν. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε το πανεπιστήμιο μια εσωτερική υπόθεση του κράτους. Η πραγματική διάσταση του πανεπιστημίου είναι διεθνούς εμβέλειας, γιατί είναι, έχουν διεθνή χαρακτήρα και τα επαγγέλματα και η έρευνα. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για προσκόμματα και ένα είδος τροχοπέδι στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης. Αυτός είναι ένας στόχος που έχει οικονομική σημασία και ανταποκρίνεται και στις νεανικές φιλοδοξίες. Ποιος θα ανταποκριθεί τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό το θέμα είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να προβάλλει μία πολιτική που να δώσει κίνητρα. Το άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας μιλά για καθήκοντα της Ένωσης και για την αναγνώριση τίτλων, για την προώθηση της ανώτατης εκπαίδευσης ως προς την ευρωπαϊκή της διάσταση. Γι' αυτό η έκθεσή μας κινείται πέραν των κρατών. Μιλάμε για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Και η συνάντηση των Υπουργών Παιδείας όπως η προσεχής που προβλέπεται στη Βουκουρέστη θα προωθήσουν αυτό, αυτή τη διάσταση του ζητήματος. Εμείς ε, μιλάμε για ε, τον βαθμιαίο χαρακτήρα για να προωθήσουμε όλες τις δραστηριότητες για να δώσουμε ευρωπαϊκό χαρακτήρα σε όλα τα πανεπιστήμια. Επίσης μιλάμε για ευελιξία το, του κορμού μαθημάτων, learning outcomes και ούτω καθεξής. Ε, ε, αποτίμηση της ποιότητας και ούτω καθεξής για να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων ακαδημαϊκών σχολών. Και στο τέλος να φτάσουμε σε αυτόνομες διαδικασίες. Να άρουμε τα κοινωνικά προσκόμματα για τους ε, πιο φτωχούς φοιτητές. Να αλλάξει η διδακτική μέθοδος, να είναι learning centered, να προωθήσουμε την ανώτατη εκπαίδευση γενικότερα ε, επικεντρώνοντάς την στην επιστήμη. 900 χρόνια πριν στη Μπολόνια ο Νέριο μίλησε για την Alma Mater και μίλησε για την Ένωση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Τότε δεν υπήρχαν κράτη. Σήμερα που υπάρχουν κράτη υπάρχει ένας έντονος κρατισμός. Γι' αυτό θα θέλαμε να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Ιθαγένεια. Ευχαριστώ. Έχουμε πέντε συναδέλφους που έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο και ξεκινάμε με την κυρία Ραόιτοβα. Ευχαριστώ. Ε, βλέπουμε ότι οι περικοπές στους πόρους για την εκπαίδευση ε, είναι πολύ δυσμενείς διότι τα κράτη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 3% του ΑΕΠ στην ε, εκπαίδευση για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να εμπλακούν ε, περισσότερο εις το τομέα της εκπαιδεύσεως παρόλη την κρίση γιατί διαφορετικά θεωρητικά θα καταλήξουμε με εκατομμύρια ανέργους πρέπει να αυξηθεί η κινητικότητα να υπάρχει αναγνώριση των διπλωμάτων και μία σύγκληση ε, των προγραμμάτων ε, εκπαιδεύσεως χαιρετίζω αυτή την έκθεση η οποία τονίζει και τις ε, αδυναμίες της διαδικασίας της Μολόνια που θα έπρεπε να επιτρέψει να επανέλθουμε εις την ε, πρόοδο. Ο κύριος Κάιτσιν έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπερλινκουέρ για τη θαυμάσια έκθεσή του. Η αναγνώριση των διπλωμάτων ευτυχώς σε πολλές χώρες είναι μια αργή και δαπανηρή διαδικασία δυστυχώς. Εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να περιορίσουμε την ανεργία, και να αξιοποιήσουμε την κινητικότητα των νέων πρέπει να καταργήσουμε τον προστατευτισμό που εξακολουθεί να ισχύει σε ορισμένες χώρες ως εμπόδιο για τα μηβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να προβάλλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο δύο θέματα τουλάχιστον. Την, την ε, ε, ε, αντιστοιχεία των διπλωμάτων και η νομοθεσία που θα διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και των πτυχίων σε επίπεδο bachelor ή masters. Αν δεν το κάνουμε αυτά σε υπερεθνικό επίπεδο θα εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε προστατευτισμό στην παιδεία. Ευχαριστώ κύριος Μιγκάλης και έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα σαν ομάδα για την ψηφοφορία. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στο κείμενο που είναι καλά η αναγνώριση των προσόντων παραδείγματος χάρη και μας ενδιαφέρει επίσης η συνεργασία με τις τρίτες χώρες στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και τα υποστηρίζουμε, αλλά υπάρχουν και κάποια σημεία που μας προβληματίζουν. Ο εισηγητής έλεγε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους φτωχότερους για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν, να μορφωθούν. Ταυτόχρονα μιλάμε για μία υποχρεωτική περίοδο ε, σπουδών αλλά αυτό θα αυξήσει το κόστος υπερβολικά. Δεν υπάρχει ομοιογένεια σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ο Πιότρ Μπόρις έχει το λόγο. Θα ήθελα να ε, μιλάμε εδώ και καιρό και πολλά χρόνια για τη διαδικασία της Μπολόνια σωστό είναι να την αξιολογήσουμε αλλά τι στοχεύουμε αυξημένη κινητικότητα των φοιτητών μας εφόσον έχουμε μια ανοιχτή αγορά εργασίας και είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και υπάρχουν χιλιάδες χιλιάδες παραδείγματα πολωνών φοιτητών που βρίσκονται στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη σε αυτή την κινητικότητα των νέων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διασύνδεση ανάμεσα στο Εράσμου, στην αμοιβή γνώση των διπλωμάτων και τη διαδικασία της Μπολόνια αφετέρου. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία της Μπολόνια θα ε, προωθηθεί συστηματικά δεν, μπορούμε να συγκρίνουμε όλα τα πανεπιστήμια στο ίδιο επίπεδο όπως παραδείγματο χάρη μουσικές ακαδημίες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει διαρκής παρακολούθηση της ε, διαδικασίας της Μπολόνια. Η Σύνοδος για τη διαδικασία της Μπολόνια που θα καθορίσει τις προτεραιότητες για τα τρία επόμενα χρόνια. Κύριος στόχος της διαδικασία της Μπολόνια, μην το ξεχνάμε, είναι η προϋπόθεση ότι κάθε φοιτητής του ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου έχει... να έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις σπουδές του ώστε να αποκτήσει τα αναγκαία προσόντα τα οποία και θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δούμε πόσα πανεπιστήμια μπορούν πράγματι να προσφέρουν παιδεία, ε, μόρφωση υψηλής ποιότητας. Τα κονδύλια που μπορούμε να επενδύσουμε στην παιδεία είναι περιορισμένα. Θα έπρεπε λοιπόν να εστιάζονται σε μέτρα που θα προωθήσουν την ποιότητα. Τέτοιες σχολές, και, τα, και τις σχολές και τα πανεπιστήμια που μπορούν να προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης είναι κάτι το σημαντικό ώστε να εκδίδουν ε, ε, διπλώματα τα οποία γίνονται παντού, να αναγνωρίζονται παντού. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τώρα την κυρία Βασιλείου να παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή τον κύριο Μπελίνγκουρ για την πολύ επίκαιρη έκθεσή του. Ολοκληρώσατε το έργο σας πολύ αποτελεσματικά καθώς προετοιμαζόμαστε για την Υπουργική Σύνοδο της Μπολόνια στην οποία αναφέρθηκαν πολλοί ομιλητές. Ευρωπαϊκός χώρος της τριτροβάθμιας εκπαίδευσης χρήζει δημόσιας, της δημόσιας προσοχής που έχει εξασφαλίσει σήμερα. Η διάσκεψη της Μπολόνια θα λάβει χώρα σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη με ανεργία μεταξύ των νέων ειδικότερα που έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά επίπεδα σε πολλές περιοχές της Υπήρου μας. Είναι λοιπόν αυτή η κατάλληλη στιγμή να ζητήσουμε πώ η διαδικασία της Μπολόνια για την τριτο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να μας βοηθήσει να αναζητήσουμε λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και αποτελεί όμως και μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε την πρόοδο μετά από μια δεκαετία εκθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτή την έκθεση που υπογραμμίζει τα κύρια επιτεύγματα της διαδικασίας της Μπολόνια μέχρι σήμερα και δείχνει την οδό που πρέπει να ακολουθήσουμε για το μέλλον. Πρόκειται για ουσιαστική συμβολή στη συζήτηση, σημαντική αυτή συζήτηση για το μέλλον της αυτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Έχουμε, έχουν σημειωθεί ουσιαστικές πρόοδες στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια. Δύο τρίτα περίπου των 47 συμμετεχουσών χωρών έχουν πάνω από 90% των προγραμμάτων σου να έχουν ευθυγραμμιστεί με το σύστημα των δύο κύκλων της Μπολόνια. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει αυξηθεί και η διασφάλιση ποιότητας έχει επίσης βελτιωθεί. Και όμως ε, ε, ε, μας περιμένουν πολλές άλλες προκλήσεις. Η συγκρίσιμη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς των Πιστοτικών Μονάδων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης και η διαφανής εφαρμογή των πλαισίων για τα προσόντα είναι μεταξύ των σημαντικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση ε, της ποιότητας, για την ε, πρόθεση της κινητικότητας, εξασφαλίζοντας ότι τα συστήματα και τα προγράμματά μας θα, έχουν, θα είναι πιο σχετικά για τις αγορές εργασίας. Τέλος, πρέπει να ανοίξουμε την πρόσβαση ώστε μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών από οποιαδήποτε προέλευση να μπορούν να απολαύσουν των ωφελο... ωφελημάτων της ε, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της σε στενή συνεργασία με όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στην εργασία της Μπολόνια για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να τονίσω την ε, δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα και ιδίως το γεγονός